Herr Präsident! Αξιότιμοι κυρίε και κύριοι, παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσουμε και πάλι την συνεδρίαση. Έχει εγκριθεί το η χθεσινή μερίσια διάταξη και είναι διαθέσιμο. Υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις, δεν ισχύει αυτό, άρα εγκρίνεται Εγκρίνονται τα πρακτικά. Πάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ε, πρόκειται